μείωση θα επηρεάσει αυτές τις ομάδες. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της προσοχής, της μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση. Και ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο σε σχέση και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μάλκολμ Χάρμπουρ, για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Πρόεδρε, να περιμένουμε ένα λεπτό για να έρθει ο κύριος Μπαρνιέ, πριν ξεκινήσω. Félicitations. Mr. President, it's a privilege. Κύριε Πρόεδρε, είναι προνόμιο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να είναι σε θέση να καλωσορίσει για πρώτη φορά το καινούριο μας Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και έχουν επέλθει πολλές αλλαγές γιατί μέσα σε δύο μέρες από την έδρα του στα πίσω έδρανα έχει έρθει στην πρώτη σειρά εδώ. Συγχαρητήρια κύριε Επίτροπε. Η Επιτροπή μας είχε την ε, ευκαιρία αναφορικά με το θέμα αυτό να διευθετήσει κάποια πράγματα και να εκφράσει τις ανησυχίες της για τις εξελίξεις σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Έχουν προκύψει διάφορες ασάφειες ως προς το συνολικό νομοθετικό καθεστώς για τα τυχερά παιχνίδια στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Σίγουρα, Επίτρεπε, ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα Ελπίζουμε όμως να το θέσετε και ως θέμα υψηλής προτεραιότητας, γιατί η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε διενεργήσει δικές μας μελέτες, δικές μας ε, εκθέσεις, έχουμε συντάξει ίδιες πρωτοβουλίες και άλλοι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο αργότερα. Ε, θέλω να ξέρετε ότι το ενδιαφέρον μας παραμένει αμύωτο για το θέμα αυτό και θα γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι και σε επίπεδο Συμβουλίου συναντώνται και συνέρχονται τα κράτη-μέλη σε τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, διότι αυξάνονται τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο σε σχέση με ό,τι γίνεται στο εσωτερικό των κρατών μελών. Το θέμα αυτό δεν προϋποθέτει νέα απελευθέρωση των αγορών ε, τυχερών παιχνιδιών, ούτε απαραίτητο αναλαμβάνεται νέα πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι η αυξημένη δημοφιλία των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο ουσιαστικά πιέζει προς τα κάτω διάφορα κρατικά μονοπόλια και υφιστάμενους φορείς διενέργειας τεχνικών παιχνιδιών οι οποίοι κατά κύριο λόγο ελέγχονται από τα κράτη και αποτελούν πολύ μεγάλο πόρο εισοδημάτων για τα ίδια τα κράτη-μέλη. Από εκεί και πέρα, πολλές ε, υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ορισμένοι συνάδελφοι ίσω αναφερθούν σε αυτές. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Ωστόσο, ε, σύμφωνα με τη δική μας ε, οπτική γωνία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες ενίοτε παρουσιάζουν ασυνέπεια μεταξύ τους και αυτό δεν βοηθά καθόλου την κατάσταση αντιθέτω την περιπλέκει έτη περαιτέρω. Και θα γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει και διάφορε διαδικασίε επί παραβάση για θέματα τυχερών παιχνιδιών, όχι απαραίτητα τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, τίθεται το θέμα κατά πόσο ένα φορέα εκμετάλλευση μια εταιρεία μπορεί να πάει και να εγκατασταθεί από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Όλα αυτά δείχνουν ότι η χρονική συγκυρία είναι η απολύτως κατάλληλη ώστε να, για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασχοληθεί με τις διαδικασίες επί να εξετάσει τις αποφάσεις που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να χαράξει μια στρατηγική, προτάσεις για το πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε και να διορθώσει ενίοτε και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις ασυνέπειες. Διότι και από πλευράς καταναλωτή θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και από πλευράς νομοθέτη θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ρύθμιση. Μπορούν να ρυθμιστούν αυτές οι αγορές και Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και οργανώνουν τυχερά παιχνίδια είναι διαθέσιμες και είναι δεσμευμένες να ε, ε, επιβάλλουν και να εφαρμόζουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να τηρούν όλες τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις. Πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Είναι θέμα και προστασία του καταναλωτή, αλλά και θέμα που έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να σεβόμαστε του πολίτε μα και να σεβαστούμε το γεγονό ότι πολλοί θέλουν να έχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι κανεί θέλει να το απαγορεύσει αυτό. Άλλωστε και στην πράξη θα ήταν αυτό ανεφάρμοστο η απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται να συμμετάσχει κανείς σε τυχερό παιχνίδι στο διαδίκτυο που οργανώνεται από εταιρεία που δεν έχει έδρα στο δικό του κράτος μέλος και αυτό δεν μπορεί να γίνει επιτρεπτό. Ένας Βρετανός πολίτης ο οποίος ας πούμε παίζει λότο στο διαδίκτυο το οποίο οργανώνεται από τη Βρετανική Υπηρεσία Λότο αλλά αν μπει στο διαδίκτυο από την Ισπανία και κερδίσει είναι παράνομο ο Βρετανικός Φορέας Διοργάνωσης του Λότο να τον πληρώσει, να του δώσει τα κέρδη του στην Ισπανία. Είναι περίπλοκο λοιπόν το θέμα. Όλοι οι συνάδελφοι θα συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση πολύ επικοδομητικά. Πρέπει όμως και εσείς, Επίτροπε, να θέσετε το θέμα αυτό υψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων σας. Σας ευχαριστούμε. Σας καλωσορίζουμε και πάλι, ε, κύριε Επίτροπε, στο Σώμα των Επιτρόπων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτέ. Αντιλαμβάνεστε ε, πόσο χαίρομαι που σας βρίσκω 48 ώρες μετά την εκλογή ε, και ε, επικύρωση του Κολεγίου των Επιτρόπων σχετικά με την ε, ε, νέα εργασία μου για την προστασία των καταναλωτών και την εσωτερική αγορά. Ε, διαφορετική τοποθέτηση αλλά το ίδιο πνεύμα. Και θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα διότι όπως είπατε η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μία διαδικασία σε σχετικά με ε, ε, τα διασυνοριακά στοιχήματα διότι η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν προτείνει αλλαγές στην εθνική νομοθεσία για να ανταποκριθούν στη διαδικασία παραβίασης. Θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία παραβίασης αλλά η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα χειριστεί αυτούς τους φακέλους. Υπάρχει και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην περίπτωση της Πρωτογαλίας όπου υπάρχει ένα εθνικό μονοπόλιο το κρατικό το οποίο ελέγχει στενά τα τυχερά παιχνίδια και ε, δεν ε, ε, θα αλλάξει βέβαια το γεγονός αυτό της διαδικασίας παραβίασης διότι οι περιπτώσεις εξετάζονται βάσει των, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Τέτοιοι περιορισμοί λοιπόν θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει του γενικού συμφέροντος και δεύτερον να είναι αναλογικοί σχετικά με τις ανάγκες οι οποίες θα, τους περιορισμούς οι οποίοι θα εφαρμόζονται όπου είναι αναγκαίο. Θα χρειάζεται όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να δώσει στα κράτη-μέλη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις όποτε το θεωρούν ε, αναγκαίο βάσει των ε, προδιαγραφών. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλεί εναλλακτική πρακτικές λύσεις στις διαδικασίες παραβίασης. Θέλω να ξεκινήσω μία επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη επί τούτου, διότι δεν υπήρχε διαβούλευση των κρατών μελών επ' αυτού από, από όταν τα κράτη-μέλη αποφάσισαν το 2006 να αποσύρουν τα τυχερά παιχνίδια από την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θα παρακολουθήσω το θέμα θέμα και το Κοινοβούλιο με την πρωτοβουλία της κυρίας Σάλτερ Μόζε στις 10 Μαρτίου υιοθέτησε μία έκθεση παρόλο που παρουσιάζεται μία αντιπρόταση. Θεωρώ ότι η πρότασή σας είναι καλό σημείο εκκίνησης για να επιλύσουμε αυτό το περίπλοκο θέμα, να εξετάσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους τα κράτη-μέλη περιορίζουν τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και πρέπει επίσης να εξετάσουμε εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην κοινωνία και ιδίως στον εθισμό στα ταχερά παιχνίδια. Ε, όπως σας είπα ξεκινήσαμε πριν από δύο μέρες, δεν έχουμε ακόμη ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί. Θα ακολουθήσω με μεγάλη προσοχή ό,τι έχετε να μου πείτε σήμερα και θα εξετάσω διάφορες υποθετικές λύσεις, δηλαδή την πράσινη βίβλο επί του θέματος. Σας ευχαριστώ και πάλι και ε, ε, για την ε, συνδρομή σας και για τις εργασίες και τη βοήθειά σας στην Επιτροπή τις οποίες θα αναλάβω. Κύριο Σβάμπ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν εν ονόματι του ΕΛΚ θα ήθελα να σας ε, εκφράσω τη χαρά μου διότι κύριε Επίτροπε ε, μας είπατε ότι θα εξετάσετε τους, τα θέματα εστιασμένα και θα προωθήσετε το θέμα στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου σχετικά με την, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο διότι αυτό είναι το θέμα μας σήμερα και θα ήθελα να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε στην απόφασή του προς τα κράτη-μέλη ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μία αγορά σαν τις άλλες παρόλα αυτά όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει κοινοτικά να συμφωνήσουν επί ενιαίων κανόνων και αυτή η προσπάθεια του Συμβουλίου μέχρι στιγμής δεν έχει εξαχθεί επικοδομητικά και γι' αυτό νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή από κοινού πρέπει να προχωρήσουν με κριτικές ερωτήσεις και να προωθήσουν το θέμα. Και εδώ αναφέρομαι στην εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών διότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν με πείθουν. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας λέγεται ότι σε περίπτωση τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο τα κράτη-μέλη μόνα τους μπορούν να εφαρμόσουν στόχους για τους καταναλωτές και να καταπολεμήσουν μόνα τους την ε, εγκληματικότητα. Αλλά κυρίες και κύριοι βλέπετε ότι όταν ε, υπάρχουν ριζικές ε, εγκληματικές πράξεις μέσω του διαδικτύου η Ευρώπη δεν θα έχει καμία δυνατότητα να επιζητήσει λύσεις και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να προχωρήσει και ο μόνος τρόπος να υπάρξει λύση θα είναι ε, να επιζητηθεί αυτή ε, διασυνοριακά όπου ε, οι χώρες θα κρατήσουν τις παραδοσιακές δομές τους αλλά όπου οι καταναλωτές θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ ώρα για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε που δεν με ικανοποιούν πλήρως, αλλά για να ξεκινήσω από την αρχή. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο, την απελευθέρωση την αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε επανελάμβανε ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιληθεί το θέμα και γι' αυτό δεν πρέπει τα κρατη αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ρυθμίσουν τα τυχερά παιχνίδια και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική οδηγία αφαίρεσε από την οδηγία υπηρεσιών τα τυχερά παιχνίδια για να υπάρχει ένας φραγμός και προστασία για τους πολίτες για να περιορίσουμε την εγκληματικότητα αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι πάντοτε όποτε προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χάνει και αυτό πρέπει να το παραδεχθείτε και ελπίζω κύριε Μπανιέ ότι θα εφαρμόσετε αυτό που είπατε δηλαδή ότι θα βρείτε μια διαφορετική λύση σε αυτόν τον τρόπο διότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή τη μεθοδολογία. Και πρέπει να σας πω ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πολύ συνεπείς. Πάντοτε διευκρινίζουν ότι τα κράτη-μέρη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες κατά τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών ε, και να μπορεί να ελέγχεται και η προστασία κατά της εγκληματικότητας. Δεν είναι υποχρεωμένα να ανοίξουν αυτή την αγορά δεν είναι υποχρεωμένοι να επιτρέψουν το κομμάτι αγοράς από τρίτες χώρες ε, και θα πρέπει ε, να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι οι οποίοι θα είναι αποτελεσματικοί. Αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να το καταλάβει και να λειτουργήσει ε, αρμοδίως. Αυτό όμως πρέπει να οδηγήσει σε σκέψεις για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο που δεν υπάρχουν σύνορα και όπου υπάρχουν σαφές, σαφείς προσβάσεις των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους ελέγχους, τους κανόνες σε αυτό το τομέα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους πολίτες και να τους σεβόμαστε. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κρόιτσμαν για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, όταν ε, ε, ζητούμε να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ισχύσουν και ενιαίοι κανόνες και το θέμα των τυχερών παιχνιδιών έχει τρεις πτυχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, δηλαδή θα, πώς μπορούμε καλύτερα να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, πώς μπορούμε καλύτερα να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα και να αποτρέψουμε τις παράνομες πράξεις ε, στα θέματα αυτά ε, είδαμε πώς λειτουργούμε στο θέμα των τυχερών ε, παιχνιδιών. Η απόφαση του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφανίζει τη θέση του και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιλύσουν το θέμα ε, εθνικά. Δηλαδή ε, η εθνική αντιμετώπιση είναι η καλύτερη για να αντιμετωπίσει κανείς ε, τη διαφθορά. Αλλά πιστεύω ότι όντως πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτά τα θέματα εις εθνικό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν όλα τα θέματα να ρυθμιστούν βάσει της ενιαίας αγοράς ιδίως όταν πρόκειται για νέους και για εθισμένους στα τυχερά παιχνίδια. Καλύτερα να αποφύγουμε ε, και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο διαδίκτυο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει σωστός έλεγχος για να μπορέσει κανείς να ρυθμίσει τα βασικότερα θέματα που αφορούν τους πολίτες διασυνοριακά να χρηματοδοτήσουμε τα πολιτισμικά θέματα και να μην νομιμοποιήσουμε τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα ε, διότι ε, θα πρέπει αυτά να καταπολεμηθούν ε, και όσον αφορά την χρήση τυχερών παιχνιδών στο διαδίκτυο θεωρώ ότι πρέπει να καλύψουμε το κενό που έχει δημιουργηθεί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η επιτήρηση της αγοράς είναι το, η λέξη κλειδί. Εάν συμφωνήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα κράτη-μέλη βάσει της αρχής της επικουρικότητας έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σύμφωνα με τις παραδόσεις τους στον τομέα, τότε θα υπάρχει πιο αποτελεσματικός έλεγχος και καλύτερη υποπτία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε τώρα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ και ε, μετά ε, δεν έχω πολλά να πω μετά από τους προλαλήσαντες αλλά σαν πολιτική ομάδα πρέπει να σας πω ότι στηρίζουμε πλήρως το ψήφισμα το οποίο υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ε, ε, θεωρούμε ότι ε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν πολύ σαφής και όχι αμφίσιμη και θα ήθελα να προσθέσω ότι η διαβούλευση είναι καλύτερη από τις διαδικασίες κυρώσεων να λάβουμε υπόψη τις εθνικές ιδιομορφίες και να λύσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Um, Κύριο Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μιλώ ως πρώην υπουργό υπεύθυνο για τα τυχερά παιχνίδια στη Βρετανία. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη του ελεύθερου εμπορίου, η οποία είναι αντίθετη στον προστατευτισμό που καταστρέφει τα εμπόδια εμπορίου, τα υποστηρίζω. Και κάποιοι από αυτούς που ζητούν ανοιχτή Ευρώπη είναι αυτοί που υποστηρίζουν και τα μονοπόλια των τυχερών παιχνιδιών. Τα μονοπόλια ελέγχουν πολύ καλύτερα τα τυχερά παιχνίδια. Πάντως τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν αυτά τα επιχειρήματα. Περισσότερο άλλαγχο και περισσότερα χρήματα για τι εθνικέ κυβερνήσει οδηγούν μόνο αυτά τα μονοπόλια. Δεν είναι αυτό η ανοιχτή, διαφανή Ευρώπη που θέλω. Που λέει κάνε ό,τι θέλω, όχι ό,τι κάνω. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον προστατευτισμό σε μια, ένα κράτος μέλος. Μια ανοιχτή αγορά μπορεί να δώσει μια ισοδύναμη προστασία των πολιτών όπως και κάθε σωστά ελεγχόμενο μονοπόλιο. Και συνεχώς έχουμε και αποφάσεις του ΔΕΚ. Ίσως το έχουν βαρεθεί αυτό στο Λουξεμβούργο. Αλλά υπάρχει επίσης και τρομερή σιωπή της Κομισιόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι τώρα να αναλάβουμε δράση. Δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω νομική αβεβαιότητα το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει σημάδι ότι θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα και ένα μήνυμα στο Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε. Με τη νέα Κομισιόν αναμένουμε μια νέα όθηση. Έχω, ελπίζω πολλά από σας, Επίτροπε Μπαρνιέ, να ακούσετε τις συμβουλές που ακούτε και να βρείτε μια στρατηγική ότι τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο θα είναι τμήμα της εσιαίας αγοράς με την κατάλληλη βεβαίως ρύθμιση. Ευχαριστούμε ο κύριος Jong. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα τυχερά παιχνίδια υπάρχουν και στην Ολλανδία βεβαίως. Όμως είναι ελάχιστες οι πιθανότητες κέρδους. Πάντως το όλο, όλη αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες στις κάτω χώρες υπάρχει μια νομοθεσία η οποία ελέγχει τα τυχερά παιχνίδια και πρέπει ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη τους νέους. Οι νέοι τώρα έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εδώ δεν μιλάμε για ενιαία αγορά. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Κατά την άποψή μου το προφορικό ερώτημα το οποίο οδήγησε στη συζήτησή μας δεν θίγει την καραδιά του προβλήματος. Νομίζω ότι με το όρο διαδίκτυο δεν μιλάμε, μόνο, δεν μιλάμε εδώ για υπεύθυνη ε, άσκηση των τυχερών παιχνιδιών. Πρέπει να απαγορευθούν τέτοιου είδους παιχνίδια. Καλό λοιπόν την Κομισιόν να μην κάνει καμία πρόταση ρύθμιση για την μείωση της προστασίας των καταναλωτών. Το αντίθετο μας χρειάζεται. Χρειάζεται επαρκές επίπεδο ρύθμισης και να μην προσφεύγουμε συνεχώς στο ΔΕΚ αλλά να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Ο κύριος Πάσκα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 Σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια θα ήθελα να σας πω ότι βλέπω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μία ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ελεύθερη ε, προσχώρηση προς το διαδίκτυο και για τους νέους και για τα παιδιά ε, και η ευθύνη ε, για τα ε, τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο πρέπει να επιβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος θα αναλάβει αυτή την θα αναλάβει αυτή την ευθύνη οι γονείς δεν είναι δυνατόν εμείς σαν ευρωβουλευτές μπορούμε να νομοθετήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο και από εκεί και πέρα να υπάρχει μία εφαρμογή η οποία θα εξασφαλίσει ε, την προστασία των παιδιών. Διότι πρέπει όπως και στον τομέα της πορνογραφίας να δράσουμε επειδή οι γονείς δεν μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βουλίο φέρουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο. Εμείς ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ιδίως τους ψηφοφόρους μας. Επίσης όσον αφορά την, ε, τον έλεγχο των χρημάτων, ε, των χρηματικών κερδών διότι, ή των χρηματικών κυρώσεων, διότι οι κυρώσεις, οι χρηματικές που επιβάλλονται θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ε, ε, για την ε, ε, ε, ε, για την επιμόρφωση, για πολιτιστικά θέματα και εγώ σας ρωτώ χρησιμοποιούμε τα χρήματα αυτά για τον αθλητισμό οι παίκτες στο διαδίκτυο των τυχερών παιχνιδιών δεν θα στραφούν σε άλλες μεθόδους θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε καταρχήν να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των παιδιών συγχρόνως όμως να μην χάνουμε τους σπόρους ε, οι οποίοι διατίθενται στα τυχερά παιχνίδια. Ευχαριστώ η κυρία Ρόιτοβα τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί και έτσι πολλοί παρακάμπτουν την εθνική νομοθεσία. Παραμένει όμως το ερωτηματικό ως προς το κρατικό μονοπόλιο για τη διοργάνωση ε, στοιχήματος. Είναι κάτι που αφορά άμεσα και τους νέους. Το IGC αναγνωρίζει ότι λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θέσουν περιορισμούς. Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο δεν γνωρίζουν σύνορα. Και κάθε χώρα έχει δική της νομοθεσία, διαφορετική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Δεν αρκεί να παρακολουθούμε μόνο την κατάσταση, να παρακολουθούμε την ποιότητα δηλαδή, θα πρέπει να διενεργούμε και αποτελεσματικούς ελέγχους και μάλιστα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό και ζητήσαμε από την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση κανονισμού για το διαδικτυακό στίχημα και τα λοιπά τυχερά παιχνίδια. Διότι πολύ συχνά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο στοχεύουν κυρίως στους νέους και διαφημίζονται τα μάλα στους νέους. Είναι ένα θέμα που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, διότι δεν υπάρχουν περιορισμοί και στις διαφημίσεις. Και ε, επιτρέπονται επίσης ε, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις για διαδικτυακό στοιχημά κοντά και σε σχολεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σαντεμός. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Χαίρομαι διότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό με εσάς. Είχε διενεργηθεί μια κρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχατε εσείς τότε επιμείνει στο γεγονός ότι η εσωτερική αγορά υφίσταται προς όφελο του πολίτη και όχι το αντίθετο. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το εφαρμόσουμε αυτό. Στηρίζω λοιπόν την πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε. Είναι κάπως ασαφής, ωστόσο είναι λογικό να υπάρξει πράσινη βίβλος για την προκειμένου μάλλον να έχουμε περισσότερα στοιχεία και να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χρειάζεται να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Υπενθυμίζω όμως ότι πράγματι το Μάρτιο ε, εγκρίθηκε η έκθεσή μου και υπήρχε γνώμη της ε, μειοψηφία, ωστόσο η ισχυρή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στήριξε την έκθεσή μου και στη συνέχεια ε, και στο Συμβούλιο πολλοί είναι υπέρ του ξεκαθαρίσματος του τοπίου Πολλοί είναι υπέρ να ρυθμίσουν καλά τα κράτη-μέλη όλο αυτό τον κλάδο του στοιχήματος ή των τυχερών παιχνιδιών. Θα πρέπει να προστατέψουμε τον πολίτη και να λάβουμε υπόψη μας και το κοινωνικό κόστος όλων αυτών των παιχνίων. Θα ήθελα όμως μια πιο σαφή απάντηση στο εξή ερώτημα. Θέση η θέση σας έχει ως στόχο να περιορίσετε τους περιορισμούς, να μειώσετε τους περιορισμούς που υπάρχουν για το θέμα αυτό για να σταματήσουμε να παραπέμπουμε τις διάφορες υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να μην παίρνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολιτικές αποφάσεις. Θα ήθελα μια σαφή απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος Έλβορντ, Είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημα για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και τα προβλήματα όταν παίζουν ανήλικοι ή ευάλωτοι καταναλωτές. Πρέπει εδώ να δείξουμε ηγετικό ρόλο και σαφή κατεύθυνση για την προστασία αυτών των καταναλωτών. Στην αρχή του Νοεμβρίου πέρυσι έθεσα το ερώτημα στην Κομισιόν και η απάντηση που έλεγα ήταν ότι η Κομισιόν είναι υπέρ πιο ασφαλών ιστοτόπων και πληροφόρησης των καταναλωτών. Επίσης ενημέρωσης προς, τον, προς τους γονείς για το τι μπορεί να συμβεί όταν είναι στο διαδίκτυο τα παιδιά τους, ιδιαίτερα για τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό πάντως το πρόβλημα είναι κρυμμένο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλιστεί ότι είναι ενήλικος όποιος παίζει. Μπορεί κανένας να παρακάμψει τις συνθήκες ασφαλείας των ιστοτόπων αυτών. Μπορεί να κλέψει πιστοτικές κάρτες ή να ε, δώσει ψεύτικη ταυτότητα. Οι εμπειρογνώμονες δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δρούν ενστικτοδός και δεν είναι οι παραδοσιακοί παίκτες που χρησιμοποιούν τα τύχερα παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιος πραγματικά παίζει γιατί χρειάζονται πόροι για να βρούμε κανένας ποιος πληρώνει, ποιος παίζει και ποιος έχει το πρόβλημα. Χρειάζονται μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τους ανηλίκους που παίζουν στο διαδίκτυο και να προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες. Κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, οι κάτω χώρες έχουν περίπου 120.000 άτομα, άτομα που είναι θυσμένα στο παιχνίδι, στα τυχερά παιχνίδια. Είναι το 1% του πληθυσμού. Αυτό οδηγεί σε κοινωνικά προβλήματα, κατεστραμμένες οικογένειες, οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα στοιχήματα, τα τυχερά παίγνια και οι συνέπειές τους να καταπολεμηθούν όσο γίνεται πιο στεναρά. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ οργανωμένη αγορά τυχερών παιχνίων. Η αγορά αυτή είναι τμήμα της εσωτερικής αγοράς και κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να την περιορίσουμε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι παράλογο. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να διευκολύνουν μια αγορά που δημιουργεί κοινωνικές δυστυχίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντισταθούν στην ελκυστικότητα των τυχερών παιχνιδιών. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει λάβει κάποια μέτρα και προβλέπει κρατικό μονοπόλιο για τα τυχερά παιχνίδια. Θα ήταν καλύτερα να μην δούμε νέα καζίνο στην Ευρώπη. Τελικά, πάντως τα καζίνο είναι το μη χείρον βέλτιστον. Τα κράτη-μέλη που επιτρέπουν τα τυχερά παιχνίδια θα πρέπει απαραίτητο να εξασφαλίσουν ότι θα αποθαρρυνθεί η αγορά αυτή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Η ερώτηση έμεσα καλή για τη δημιουργία κοινοτικής νομοθεσίας. Από τη στιγμή όμως που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέτει τα όρια και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν τα κρατη από μόνα τους, μέσα από τις εθνικές τους νομοθεσίες, να ορίζουν το πώς ελέγχεται το διαδικτυακό στίχημα, δεν υπάρχει λόγος να ζητείται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πέραν τούτου, το δικαστήριο έχει αποφανθεί στην απόφαση Schindler ότι τα τυχερά παιχνίδια έχουν ορισμένες ηθικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές εν ενέχουν υψηλό κίνδυνο παρανομίας ή απάτης και μπορούν να έχουν βλαπτικές συνέπειες στο άτομο και στην κοινωνία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αγαπητοί συνάδελφοι για αυτούς ακριβώς τους λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει ο τομέας να παραμείνει στον έλεγχο των κρατών μελών που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες τους και πώς να τις χειριστούν. Εξάλλου, αυτό υποστηρίχθηκε τόσο από τη μελέτη την οποία εκπώνησε για λογαριασμό της Επιτροπής η Swiss Institute of Comparative Law, όσο και από τη σχετική έκθεση του 2009 με εισηγήτρια τη συνάδελφο Σαρτεμόζε και η οποία υπερψηφίστηκε σε αυτό το σώμα. Αυτή η έκθεση καταλήγει ότι μια προσέγγιση αποκλειστικά στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς δεν είναι κατάλληλη σε αυτό τον πολύ ευαίσθητο τομέα και ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το ζήτημα αυτό ξεκινώ με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η δυνατότητα κράτους μέλος να απαγορεύσει σε ιδιώτες την προσφορά παιχνιδιών στο διαδίκτυο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί αυτή η αγορά που ε, ενέχει κινδύνους για τους καταναλωτές. Εν απουσία κοινοτική εναρμόνισης για τα τυχερά παιχνίδια, κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει το δικό του επίπεδο προστασίας και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι μόνο αυτά τα μέτρα. Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασίες παραβίασης για κάποια κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων είναι και η Ιταλία γιατί παραβίασαν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπερασπίσε την ε, πορτογαλική άποψη που είναι πιο περιοριστική. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν την αρμοδιότητα να ρυθμίσει τον όλο τομέα και να εναρμονίζει τα τυχερά παιχνίδια σε κρατικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να υπερβούμε τα μεμονωμένα οικονομικά συμφόρεντα, γιατί είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και ιδιαίτερα τους ανηλίκους που είναι κυρίως τα θύματα των απατών. Ευχαριστούμε. Κορέα κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Υπάρχει εδώ μία αντίφαση ανάμεσα σε δύο καλές πολιτικές της Ένωσης. Προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από την άλλη πλευρά. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διατηρήσουν αυτονομία και νομιμότητα για να ελέγξουν τις επιχειρήσεις αυτές που δρούν στο διαδίκτυο. Είναι ένας τομέας ευαίσθητος που θίγει κοινωνικές αξίες για συμπεριφορές που οφείλονται σε εθισμό στα τυχερά παιχνίδια και παραδοσιακές εθνικές ε, συνήθειες για το πού χρησιμοποιούνται στην συνέχεια αυτά τα κονδύλια. Πάντως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χρόνια τώρα έχει μια συνεπή θέση και θα πρέπει αυτό να οδηγήσει την Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν μια πολύ πιο ρητή θέση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη για την πρόληψη του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος που χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα παιχνίδια στο διαδίκτυο και να προχωρήσει σε πραγματική προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων. Κύριε Μπαρνιέ, Ελπίζουμε ότι η νέα επιτροπή που τώρα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της θα θεωρήσει αυτό το θέμα ως προτεραιότητα των εργασιών της. Σας ευχαριστούμε. Βλάσακ, 4,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζουμε, τα τυχερά παιχνίδια τη χάνουν αυστηρών ρυθμίσεων σε πολλά κράτη-μέλη. Όμως η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά, διότι τα μεγαλύτερα καζίνο τώρα λειτουργούν διαδικτυακά. Εξελίσσονται οι τεχνολογίες, τα τεχνολογικά μέσα για το διαδικτυακό στοίχημα και τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου και οι νομοθετικές εξελίξεις καθυστερούν. Επομένως, κλήθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί επί συγκεκριμένων υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου. Και αυτό δείχνει ότι η νομολογία στο θέμα αυτό είναι και αυτή ασαφής. Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο ουσιαστικά ε, καλύπτουν μια γκρίζα περιοχή δικαίου και πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είναι τα αρμόδια για την εκχώρηση αδειών διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Ταυτοχρόνως όμως επίσης πιστεύουμε ότι η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή και στην ελεύθερη ε, κυκλοφορία αν θέλετε των υπηρεσιών, ελεύθερη προσφορά των υπηρεσιών. Ε, σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, δεν μπορεί η Τσεχία να παρεμποδίσει ξένες εταιρείες να ε, προσφέρουν αυτές τις ε, υπηρεσίες μέσα στη χώρα, ωστόσο δεν μπορεί και να δώσει άδεια σε εγχώριες επιχειρήσεις για τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα και διάφορες αντιφάσεις πέρα από το θέμα της φορολόγησης. Ευχαριστώ κυρία Εσαγιάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαγράψει μία σαφή γραμμή η οποία πρέπει να εφαρμοστεί διότι τα τυχερά ε, παιχνίδια δεν είναι μία ε, παροχή υπηρεσιών αλλά συνεπάγονται και, κοινωνικά, ε, και κοινωνικές δαπάνες. Το θέμα αυτό είναι πολύ βασικό και η εμπλοκή του Κοινοβουλίου τώρα είναι πολύ ουσιαστική διότι έχει νέες αρμοδιότητες βάσει ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Το, ε, ε, ο αθλητισμός δεν πρέπει να οδηγήσει σε ατυχερά παιχνίδια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει την συνεκτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ βασικό να μπορέσει κανείς να ε, περιοριστεί ε, τις εγκληματικές δραστηριότητες και ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε το παράδειγμα σχετικά με την Πορτογαλία. Δεν είναι όμως αναγκαία μόνο η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των κυρώσεών του, αλλά θα πρέπει υπάρχει μια ευρωπαϊκή λύση διότι κάθε κράτος αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει το οικονομικό κόστος μόνο του και θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση. Η αύξηση των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι ε, μια φυσική καταστροφή, μπορεί κανείς να τα καταπολεμήσει. Ακόμη και οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο θα πρέπει να σέβονται την νομοθεσία των κρατών μελών. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ενθαρρύνω να καταρτήσετε μία πράσινη βίβλο για τα τυχερά παιχνίδια, πράγμα το οποίο θα ε, μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τα τυχερά παιχνίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η κυρία Σίλα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ τους προηγούμενους ομιλητές για την συνεισφορά τους και τις συναδέλφους για την τεράστια προσπάθειά τους. Όπως είπαν προλαλήσαντες, το να παίζει κανένας δεν είναι μια οποιαδήποτε υπηρεσία και οι αρνητικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών δεν μπορούν παρά να υπογραμμιστούν όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο δίκτες που προσμετρούν τη σοβαρότητα. Ένας είναι ένας δείκτης για τη σοβαρότητα και την ε, σημασία και άλλος ένας καναδικός δείκτης και στη Βρετανία είπε ο Ολλανδός ότι είναι 1% του πληθυσμού επηρεάζεται αλλά στη Βρετανία είναι 236.000 άτομα που έχουν εθισμό στα τυχερά παιχνίδια. Ποιος είναι ο αριθμός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν το σκεφτείτε ε, αν τελικά εμφανιστεί αυτή η πράσινη βίβλος εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να έχει πραγματικά στατιστικά στοιχεία. Μία μελέτη για τις επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών και στο διαδίκτυο και εκτός. Είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για να ε, συζητήσουμε το θέμα και θα ήθελα να σχολιάσω και τα αποφάσεις του δικαστηρίου. Αν κοιτάξετε τι λέει, λέει για να προβλεφθεί και να παρεμποδιστεί η εγκληματική δραστηριότητα. Υπάρχουν καρτέλ και εγκληματικό ε, ε, έγκλημα που χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, να μην χρησιμοποιηθεί αυτό ως βιτρίνα για παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε με τις προσπάθειές σας και κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Δεν είναι το πιο εύκολο θέμα για να ξεκινήσετε τη θητεία σας στην Κομισιόν, αλλά ο προκάτοχός σας, ο κύριος Μαγκρίβη, σίγουρα μερικές φορές πήγαινε και έπαιζε, του αρέσανε πολύ οι κούρσες και έβαζε και κανένα στοιχηματάκι. Για το θέμα αυτό πάντως υπάρχουν εδώ δύο σκολές σκέψεις. Πάντως αυτή του Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη σύμφωνα και με το ψήφισμα του Μαρτίου πέρυσι. Καλό θα ήταν να σας διαβάσω τρεις γραμμές από αυτό το ψήφισμα που λέει τα κράτη-μέλη έχουν συμφέρον και δικαίωμα να ελέγξουν και να ρυθμίσουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών. Και ξεκάθαρα λέει ότι όσοι δρούν στο διαδίκτυο πρέπει να σέβονται την νομοθεσία των κρατών μελών όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες. Και μία προσέγγιση μόνο με βάση την ενιαία αγορά δεν είναι η κατάλληλη σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Το πρόβλημα για μας ως νομοθέτης και κράτη μέλη είναι ότι η αγορά είναι πιο μπροστά από εμά. Οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει την υφιστάμενη νομοθεσία και το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον, είτε μας αρέσει ή όχι. Ο κόσμος παίζει. Εγώ καλύτερα να αγοράζω παπούτσια. Άλλοι βεβαίως τη βρίσκουν αλλιώς. Πάντως συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα με τα τύχερα παιχνίδια είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα με όσους έχουν εθισμό και μην ξεχνάτε ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη προωθούν τα λαχεία είναι μια νόμιμη προώθηση ενός πιθανού εθισμού δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρο πού ακριβώς είναι η διαχωριστική γραμμή. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν υπάρχει συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη και παρόλα αυτά οι πολίτες μας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτός της χώρας τους και θέλουν να το κάνουν αυτό. Άρα χρειάζεται η πράσινη βίβλος, είναι μεγάλη πρόκληση για να μαζέψετε πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και υπάρχουν πολύ μεγάλο κενό στις πληροφορίες που διαθέτουμε, γι' αυτό, αυτό το κενό πρέπει να καλύψει η Κομισιόν. Ο κύριος Ρέπο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο δεν είναι μια υπηρεσία όπως οι άλλες. Ε, συνεπάγονται κοινωνικές ε, σοβαρές συνέπειες. Υπάρχει κίνδυνος δραστηριοποίησης του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει κίνδυνος ε, κατάρρευσης του ατόμου και οικονομικής κατάρρευσης αλλά και ψυχολογικής. Στη Φιλανδία το 2008 έγινε υπολογισμός και φάνηκε ότι 40.000 είναι οι εθισμένοι στον τζόγο, τον διαδικτυακό μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αν το εκθέσουμε αναλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δούμε ότι πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θυσμένοι στον τζόγο στην Ευρώπη και μάλιστα στο διαδικτυακό. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα ε, της απόφασης για το πώς θα διεργανώνεται ο διαδικτυακός τζόγος, όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες και ρύθμιση της αγοράς αυτής και εθνικούς ελέγχους. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τους πιο ευαίσθητους καταναλωτές, τις πιο ευπαθείς ομάδες που ε, διατρέχουν κινδύνους ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς και ε, εθισμού και να παρεμποδίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σαλβατόρε Ιακολίνο για δύο λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρτήρια κύριε Επίτροπα. Υπάρχει τεράστια αύξηση των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο που έχει μια κοινωνική πτυχή και χαρακτηρίζεται από την εύκολη πρόσβαση πολλών καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι κυρίως νέοι που γνωρίζουν καλύτερα την πληροφορική και το διαδίκτυο και αλλάζει η ζωή τους με τον ίδιο τον τζόγο. Υπάρχουν πάντως καταστροφικές συνέπειες και πολλές οι οικογένειες μπαίνουν σε ένα τούνελ από όπου δεν μπορούν να βγουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαρές συνέπειες γιατί δεν υπάρχει πλέον κοινωνική επαφή εξαιτίας της ύπαρξης του διαδικτύου. Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν εθισμό που γενικά δεν είναι αποδεκτή. Είναι ένα βίτσιο που ακόμα είναι κρυμμένο από την προηγούμενη εμπειρία μου ξέρω ότι είχαμε ένα ειδικό γραφείο για την υποδοχή τέτοιου είδους ασθενών. Είναι μια προσέγγιση που χρειάζεται θεραπευτική αγωγή και έρευνα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση και να φροντίσουμε ώστε όλοι οι εθισμοί να αντιμετωπιστούν. Αναφέρομαι στην ε, στα τοξικομανία, αλκοολισμό, ακόμα και το ίντερνετ, σε οποιοδήποτε εθισμό. Λυπάμαι γιατί ακόμα δεν δόθηκε απάντηση στο ερώτημα που έθεσα εγώ και άλλοι 42 συνάδελφοι και ρωτώ λοιπόν πότε η Κομισιόν θα ενδιαφερθεί και θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και άλλου είδους εθισμός πέρα του τοξικομανίας και πότε η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο. Η κυρία Ράπτη, ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο λόγος που στην Ευρώπη αισθανόμαστε ασφαλείς ο λόγος που η ευρώπη μετράει πια τόσα χρόνια ζωής είναι νομίζω το γεγονός ότι σεβάστηκε και σέβεται τις εθνικές ευαισθησίες. το συνεχές δίλημμα που έρχεται όμως και επανέρχεται αν τον πρώτο και κυριότερο λόγο τον έχει η ευρώπη ή τα κράτη μέλη είναι ταυτόχρονα και ζητούμενο και είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση των τυχερών παιχνιδιών ιδιαίτερα στο διαδίκτυο το διαδίκτυο είναι ένας χώρος συναρπαστικός αλλά ταυτοχρόνως ενέχει κινδύνους πάρα πολύ δύσκολα ελέγξιμους. παράλληλα η αρχή του ανταγωνισμού πυλώνας της εσωτερικής αγοράς δεν μπορεί να αγνοεί πρωταρχικά ζητήματα σεβασμού του εθνικού δημόσιου συμφέροντος. το ζητούμενο αυτής της ισορροπίας νομίζω ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις δύο αποφάσεις του δικαστηρίου που από τη μια μεριά κατανοεί και προασπίζει την έννοια του δημοσίου συμφέροντος ενώ απ' την άλλη όπως αυτή διασφαλίζεται μέσα από τις εθνικές παραδόσεις ενώ απ' την άλλη διατυπώνει ενστάσεις σε μη αναλογικά μέτρα τα οποία λειτουργούν τελικά σε βάρος του πολίτη. γνωρίζοντας τις διαβουλεύσεις που διενεργούνται αυτόν τον καιρό στο συμβούλιο περιμένουμε να ακούσουμε από την επιτροπή με ποιο τρόπο θα εργαστεί για να διασφαλίσει την εθνική αυτονομία δράσης αλλά και να δημιουργήσει μια αποτελεσματική βάση συνεργασίας ώστε να καταπολεμηθούν και το θέμα του εθισμού και το θέμα της απάτης που ενέχεται. και κλείνοντας κύριε επίτροπε να σας ευχηθώ συγχαρητήρια και να σας πω ότι εγώ πιστεύω όλα όσα λέγονται σε αυτή την αίθουσα. ακούγοντάς σας λοιπόν να λέτε ότι υπάρχει διαφορετική θέση για σας αυτή τη στιγμή αλλά το ίδιο πνεύμα περιμένω να το δω και στην πράξη. καλή δουλειά. Ο κύριος Ότμαρ Κάρας για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που σας βλέπω πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Διότι στον τομέα αυτό ε, θα ε, ανα, ασχολούμεθα με την ε, εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής. Από τη μία πλευρά χρειαζόμαστε περισσότερη εσωτερική αγορά και εφαρμογή των αρχών της εσωτερικής αγοράς, αλλά δεν θα πρέπει να μειώσουμε τις τις ευθύνες μας και θα πρέπει να δώσουμε το σήμα μας εις τα τυχερά παιχνίδια διότι όπως και στις οικονομικές αγορές και στα τυχερά παιχνίδια δεν θέλουμε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και μετά εμείς να πληρώνουμε τη λυπητερή πρόκειται για θέμα εκπαιδεύσεως πρόκειται για θέμα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος εγκληματικότητος πρόκειται για θέματα ελευθερίας στα τυχερά παιχνίδια και όλα αυτά θα πρέπει να συγκεραστούν. Δεν έχουμε έναν σταθερό ορισμό. Ε, υπάρχουν διαφορετικών ειδών τυχερά παιχνίδια, διαφορετικοί ορισμοί. Γι' αυτό και ε, χαιρετίζω την ανακοίνωση μίας πράσινης βίβλου κατά τρόπον ώστε να εξετάσουμε ε, τα διάφορα θέματα, τους διάφορους πολιτισμούς κατά τρόπον ώστε να έχουμε μία κοινή βάση. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σύγκρουση και ε, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της, να δεσμεύσει αυτά τα οποία πρέπει να δεσμεύσει και από κοινού θα πρέπει εδώ ούτε να υπονομεύσουμε το εθνικό δίκαιο αλλά αντιθέτως να υπάρξει μια ευξημένη ασφάλεια στο κοινοτικό χώρο. Ευχαριστώ κύριε Κάρας και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παντζέρη για δύο λεπτά και τριάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν στα διάφορα αριθμιστικά πλαίσια των κρατών μελών και γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ερμηνείες της νομολογίας και οδηγούν σε υψηλό επίπεδο παραβιάσεων κατά των κρατών μελών. Η απουσία ευρωπαϊκής πολιτικής δεν μπορεί να διατηρηθεί μπροστά στις προκλήσεις που μας θέτουν αυτά τα παιχνίδια η ευρεία διάδοση του ίντερνετ και το ηλεκτρονικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την προσφορά τέτοιου είδους παιχνιδιών και σε διασυνοριακό επίπεδο μάλιστα. Είμαι πεπισμένος ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κοινέ προκλήσεις για προστασία καταναλωτών και ανηλίκων, πρόληψη απατών, αλλά και την μη επιτρεπόμενη παροχή υπηρεσιών και τα κράτη-μέλη αυτό δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνο τους. Η Κομισιόν εργάζεται κατόπιν ετύπετος του Ευρωκοινοβουλίου για την επίτευξη ευρωπαϊκού πλαισίου. Αυτό είναι απαραίτητο. Δεν είναι εδώ υπό αμφισβήτηση η καλύτερη σας, η καλή σας βούληση. Καλά η πράσινη βίβλος, καλά όλα αυτά, καλή διαβούλευση. Αλλά μόνο αυτά για να βρεθεί το σωστό νομοθετικό πλαίσιο. Όχι να είναι αυτά αυτός σκοπός η Κομισιόν πολλές φορές μόνη της έχει συντάξει λευκές και πράσινες βίβλους χωρίς να αποφασίσει τίποτα. Χρειαζόμαστε αποφάσεις, όχι μόνο λόγια. Ευχαριστούμε. Κυρία Κόρολα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εάν δει κανείς τη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για θέματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, μπορεί να εξάγει τα εξής συμπεράσματα. Το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη απορρίπτουν την εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης και είναι πολύ ευαίσθητα ως προς αυτό το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Και το Δικαστήριο ε, ρητός το εξήγησε αυτό το περασμένο Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό για το Κοινοβούλιο ότι χάνει ένα από τα βασικά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει σε όλες τις διαδικασίες επί παραβάση. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τους δικούς τους στόχους για το, ε, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και να ορίσουν τα ίδια το, κράτος, το επίπεδο προστασίας που θεωρούν απαραίτητο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια. Το 2006 και το 2007 συμφώνησαν να αποκλειστεί το θέμα αυτό από την οδηγία για τα οπτικοακουστικά και από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι ε, δουλειά που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας και συνεχίστηκε μετά με την Σουηδική και την Ισπανική. Στην έκθεση σου Άλντε Μόρσε, εγώ ήμουν ε, αρμόδια για την ε, χάραξη της γραμμής από πλευράς ΕΛΚ και συμμερίζομαι την άποψη αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, Συμφωνείτε με την άποψη ότι θα πρέπει τελικά κάποια στιγμή να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθά κάπως τα κράτη-μέλη στον αγώνα τους αυτό ε, της καταπολέμησης των ε, παρανόμων ε, δραστηριοτήτων τέτοιου είδους. Και αν ναι, πώς θα το αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό, από, παρά να χρονοτριβείτε απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κύριο Σόνικ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναμφίβολα, η αγορά των τυχερών παιχνιδίων στο διαδίκτυο αναπτύσσεται δυναμικά. Το 40% ε, της αγοράς του τζόγου παγκοσμίω ε, ενυπάρχει στην Ευρώπη. Έχουν διπλασιαστεί τα ωφέλη από 6,2 σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η διαδικτυακή αγορά αναπτύσσεται, αλλάζουν οι συνήθειες των καταναλωτών και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Εάν δεν αντιδράσει, τότε για άλλη μια φορά φαίνεται ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά τους. Δεν προσφέρουν ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται σαφής ρύθμιση νομοθετική για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι απάτης, ε, νομιμοποίησης παράνομων προσόδων αλλά και αύξησης της εξάρτησης των ατόμων και του εθισμού τους στον τζόγο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί για να προστατεύσει τον Ευρωπαίο καταναλωτή έναντι των συνεπειών του διαδικτυακού τζόγου. Στο ψήφισμα του Μαρτίου αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι οι νέοι πολύ συχνά δεν είναι έτοιμοι, δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση και να καταλάβουν πως πολύ συχνά οι πιθανότητες στρέφονται σε βάρος τους και δεν έχουν τις πιθανότητες που νομίζουν ότι έχουν ε, όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, αντιδράσει καλύτερα και να ενημερώσει και η ίδια τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ξέρετε, ε, πολλά μέλη της Επιτροπής ε, όταν ήταν νέοι δεν είχαν αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, γιατί τα θέματα αυτά τότε, πριν από τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια, άνοικαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. <coughs> Σήμερα όμως είναι πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό οι Επιτροποί δεν συνειδητοποιούν το επίγον του θέματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα πρότυπα για να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ του ανταγωνισμού από τη μία και του τζόγου από την άλλη. Ε, κυρία Αντωνέσκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ για τα τυχερά παιχνίδια είτε ε, πρόκειται ε, για το διαδίκτυο είτε και κατευθείαν είναι ένα επικίνδυνο θέμα διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κέρδη και για άλλους λόγους πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να προωθηθούν τέτοιες δραστηριότητες ε, και τα κράτη-μέλη και οι Επιτροπή έχουν ένα κοινό στόχο ε, να ε, προστατεύσουν τους νέους, να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τους ε, κανόνες για την διαφήμιση και την υπερβολική χρήση στο διαδίκτυο των τυχερών παιχνιδιών, διότι διαφορετικά τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να καθορίσουν το σωστό πλαίσιο, ακόμη και αν και αν ε, δεν συμφωνούμε με την ύπαρξή τους πρέπει να πούμε ότι τα τυχερά παιχνίδια ποτέ δεν ε, ε, σέβονται τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς μόνος και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμβάλλει εις την εφαρμογή των επιταγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι από τη μία πλευρά πρέπει κανείς να συγκεράσει ε, και ε, την ε, ρύθμιση την κοινοτική και τα παράπονα των εξασκούντων αυτά τα τυχερά παιχνίδια γι' αυτό και χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία να ρυθμίσει τα τυχερά παιχνίδια και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους καταναλωτές δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι τα παιχνίδια αυτά θα μπορέσουν να διεξαχθούν αποτελεσματικά. Ο κύριος Ντότς για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο δι τον οποίον ε, ούτως ή άλλως συγχαίρω που αναλαμβάνει τις εργασίες του σαν επίτροπος. Αυτά που έχω να πω έχω να τα συνοψίσω σε τρία σημεία αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτον, σήμερα ζούμε στα, στην εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στον τομέα αυτό τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση κοινωνική και ε, οι επιπτώσεις της προκλήσεως αυτής δεν είναι, δεν είναι ακόμη πλήρως αντιληπτές. Στο ψήφισμα του 2009 είπαμε επαρκώς ότι τα τυχερά αυτά παιχνίδια μπορούν να έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις, ε, εθισμό και επιπλέον ε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι εδώ μιλάμε για κινδύνους και για τα νόμιμα τυχερά παιχνίδια ε, ε, μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάποιο ε, σκάνδαλο στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια του διαδικτύου δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν θέμα της ενιαίας αγοράς αλλά προστασίας του καταναλωτού. Αυτή είναι η πτυχή που πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλω λοιπόν να διατυπώσω δύο προτάσεις. Χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πλευρά του καταναλωτή και ε, θα ε, μπορέσει να συμβάλλει στην ε, πρόληψη του εθισμού, στην προώθηση του fair play και στο τον διαχωρισμό μεταξύ των εγκληματιών και των νομίμων παικτών. Θα πρέπει να καταρτιστούν και αξίες οι οποίες να είναι προς όλων. Η κυρία Χίγκινς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως πολλοί άλλοι τομείς και εδώ η τεχνολογία επηρεάζει αυτό τον τομέα. Γι' αυτό έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Είναι πιο εύκολο κανένας να έχει πρόσβαση και να καβάλει ένα στοίχημα. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για τα κράτη-μέλη και έχουμε περάσει όμως τώρα και σε άλλους τομείς όπου κανένας μπορεί να βάλει στίχημα Και έχουμε λοιπόν πολύ προχωρήσει στους τομείς που καλύπτουν πλέον τα τυχερά παιχνίδια. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχουν απάτες, εθισμοί. Στην Βρετανία και μόνο εκτιμάται ότι υπάρχουν 600.000 εθισμένοι που είναι μέλη του Gamblers Anonymous. Το ίδιο ισχύει και στην Ιρλανδία. Είναι κοινό το πρόβλημα στην όλη Ένωση. Α κοιτάξουμε την απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι κάθε κράτος μέλος καθορίζει δικαιού του κανόνες. Όμως εμείς χρειαζόμαστε κοινού κανόνες γιατί ο τζόκο περνάει τα σύνορα και θα πρέπει να επανέλθουμε στην εξέρεκτη σύσταση του 2009. Κοιτάξτε, τα κράτη, καλούμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να επιληθούν προβλήματα κοινωνικής τάξης εξαιτία διασυνοριακών τυχερών παιχνιδιών. Να προστατεύσουμε τους καταναλωτές κατά των απατών και χρειάζεται κοινό κανονισμό για τη διαφήμιση, προώθηση των παιχνιδιών στο διαδίκτυο και για την πίστοση. Θα πρέπει να υπάρχει μέγιστο δυνατόν ποσών για πίστοση και περιορισμούς για την ηλικία. Εδώ πολύ μιλάμε και μιλάμε για ψηφίσματα και συστάσεις, καλά όλα αυτά, αλλά στο τέλος αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν όλα αυτά δράση, αλλιώς είναι μόνο καλές προθέσεις. Μιλάμε για δράση και χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό αναμένω την απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Higgins. Η κυρία Μορκουνάιτε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κανείς δεν αρνείται το γεγονός ότι τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια δημιουργούν πολλά προβλήματα στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Οι εξαρτήσεις οξύνονται συνεχώς από το 96 και μετά. Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι μια δραστηριότητα η οποία γνωρίζει ανωδική πορεία. Και από ό,τι φαίνεται τα εξαρτημένα άτομα θα αυξηθούν, ο αριθμός τους δηλαδή. Δεν έχουμε πολλά ενημερωτικά στοιχεία για το θέμα αυτό. Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται ε, στην αγορά τη διαδικτυακή έχουν πολλούς λόγους να χαίρονται Βεβαίω οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα τη ρύθμιση των υπηρεσιών και το θέμα τη διασφάλισης ενό ελάχιστου επίπεδου προστασία. Στη Λιθουανία τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται ούτω ή άλλω. Ωστόσο, οι Λιθουανοί πολίτε έχουν πρόσβαση σε ε, τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και έτσι δεν την χάνουν τις απαιτούμενε προστασιες Εξού και είναι εξαιρετικά σημαντική η δημιουργία ενό κοινού συστήματος κοινών ρυθμίσεων με προσανατολισμένων των ρυθμίσεων αυτών στην προστασία των ανήλικων. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους όχι μόνο και όχι τόσο αν θέλετε από παιχνίδια στα οποία διακυβεύονται χρήματα αλλά κυρίως από παιχνίδια ε, τα οποία ε, δημιουργούν τον κίνδυνο απόκτησης εξάρτησης από αυτά. Υπάρχουν διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια τα οποία είναι εξαιρετικά βία και μπορεί κανείς να εξαρτηθεί παίζοντας συνέχεια στο διαδικτύο τέτοιου είδους ε, παιχνίδια. Θα πρέπει να φτάσουμε ε, σε μια ε, κοινή λύση. Όπως έχουμε τις κλιματολογικές αλλαγές, έτσι έχουμε και τις τεχνολογικές αλλαγές στο διαδίκτυο. Πρέπει να μην καθυστερούμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύγκριση. Κύριος Μπόρις, δύο λεπτά. E, Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω στην Ευρωπαϊκή να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ερώτημα. Εκ μέρους και του συναδέλφου κ. Νίτρας, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στο Στρασβούργο. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο, μπορείτε να σχολιάσετε τις πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία των κρατών μελών στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεύτερον, μήπως η Επιτροπή προβλέπει να την ανάληψη νομικής δράσης για να ρυθμίσει συναλλαγές που έχουν να κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. do końca weryfikowane i kontrolowane. w związku z tym czy zdaniem komisji ε, Θα ήθελα να ξέρω καν κατά πόσο, ε, σύμφωνα με την ε, Επιτροπή, οι κοινέ ρυθμίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υποχρεωτικέ αυτή τη στιγμή. Μια, μια όπου, σε μια συγκυρία όπου οι χώρε μέλη δεν είναι σε θέση να αναχαιτήσουν τα παιχνίδια αυτά των πολιτών πέρα από τις ε, προβλέψεις και τις διατάξεις. Έχω την εντύπωση ότι οι νομικοί κανονισμοί δεν είναι προσαρμοσμένοι στην παρούσα κατάσταση, στην αγορά που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, στην αγορά των υπηρεσιών και του Ιντερνετ. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα, τι είδου ε, δράσει προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πεδίο. Να υπάρξει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλε τι χώρε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπορή. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Μάντερ για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπαρνιέ και θα ήθελα να τον χαιρετήσω από αυτή την θέση. Η οδηγία Μπόλκενστάιν, η οδηγία για τις υπηρεσίες, την οποία συζητήσαμε Μακρόν, ε, από αυτήν αποκλείστηκαν τα τυχερά παιχνίδια, εξαιρέθηκαν τα τυχερά παιχνίδια και λυπούμε γι' αυτό. Γιατί φαίνεται ότι δεν τολμήσαμε να δούμε, να προβούμε στη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές. Προφανώς οι αρχές της χώρες μέλη έδωσαν τη, σε κάποιες χώρες έδωσαν τη δυνατότητα σε μονοπόλια. Άλλες χώρες δεν το έπραξαν. Νομίζω ότι το έδαφος εδώ είναι ιδιαίτερος ολισθηρό. Και θεωρώ ότι ο λόγος είναι η έλλειψη θάρρους να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, πολύ συχνά εφαρμόζουμε μια πολιτική στρουθοκαμιλισμού. Οι φορείς που προσφέρουν αυτά τα χερά παιχνίδια ψάχνουν τα νομικά κενά. Και η νομική εφαρμογή μέχρι στιγμής έχει προσκρούσει σε κάποια όρια αλλά η εποχή αυτή έχει παρέλθει. Χρειαζόμαστε μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τυχερά παιχνίδια. Οι πάροχοι θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, σε αυτή τη ρύθμιση, οι καταναλωτέ θα πρέπει να προστατευθούν, οι εγκληματικέ οργανώσει θα πρέπει να αποκλειστούν και να καταπολεμηθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επιτέλους να πάψουμε να επιτρέπουμε στις χώρες μέλη να διατηρούν ε, κάποια μονοπόλια ε, η περιοριστική πολιτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περιπλέκει τα πράγματα. Θα πρέπει να επιδείξουμε επιτέλους το αναγκαίο θάρρος ούτως ώστε να μερμνήσουμε για τον πολίτη και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις εγκληματικές οργανώσεις. Εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται εδώ τα τυχερά παιχνίδια ε, θα πρέπει να εμποδιστούν. Κύριε Μπανιέ, θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και ενδεχομένως θα ήταν ενδιαφέρον για σας να εξετάσετε την εφαρμογή της οδηγίας για τα τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρει ιδιαίτερως γι' αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Όμπερμαϊρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει επί της ουσίας κατά πόσο η Πορτογαλία ε, παραβάζει το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια. Η Πορτογαλία είχε απαγορεύσει σε κάποιες επιχειρήσεις να προσφέρουν τυχερά παιχνίδια online η η Επαγγελματική Ένωση της Πορτογαλίας ε, προέβαλε το επιχείρημα ότι τελικά παραβιάζεται το δικαίωμα της Πορτογαλίας για την, παροχή ελεύθερων, για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να δέχεται υπηρεσίες. Υπάρχει και μια παθητική ελευθερία των υπηρεσιών. Η χώρα επίσης δεν θα πρέπει να κάνει διακρίσεις κατά ξένων παρόχων. Ωστόσο, η οδηγία για την ελευθερία των υπηρεσιών ακριβώς θέλει να καταργήσει αυτή τη διακριτική μεταχείριση έναντι αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η ελευθερία αυτή υπαρχή υπηρεσιών μπορεί να περιοριστεί εφόσον υπάρχουν αποχρόντε λόγοι οι οποίοι απειλούν το κοινό συμφέρον. Εάν είναι αναγκαία η καταπολέμηση τη απάτη ή ο αγώνα κατά του εθισμού στα παιχνίδια αυτά. Ιδιαίτερα στο ζήτημα του εθισμού συνιστά ένα μείζον πρόβλημα, κυρίε και κύριοι. Στη Γερμανία 200.000 ε, άνθρωποι είναι επισήμω ε, εθισμένοι στα τυχερά παιχνίδια, μεταξύ αυτών και οι περισσότεροι είναι νέοι. Η ηλικία ε, τοποθετείται ήδη στα 13 που ξεκινούν. Από την άλλη γνωρίζουμε ε, αυτή την ε, προβληματική που σχετίζεται με αυστηρές ε, κυρώσεις. Τα κρατικά μονοπόλια για τα τυχερά παιχνίδια ε, δεν ε, ε, παρεμποδίζονται από τι διατάξει περί ανταγωνισμού και με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στα τυχερά παιχνίδια. Είναι μια ιδιαίτερο αντιφατική και πολύπλοκη κατάσταση και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Catch the Eye. Και ο κύριος Κολίνο έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στον κύριο Μπαρνιέ. Τις χρειάζεται τις ευχές. Ο τζόγος δημιουργεί εθισμό και επηρεάζει ολόκληρες κοινωνίες στη συμπεριφορά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ρυθμίζουν από μόνα τους τα τυχερά παιχνίδια με δικές τους νομοθεσίες. Η απόφαση για τον πορτογαλικό οργανισμό τυχερών παιχνιδιών θα επηρεάσει αρνητικά τις δυνατότητες εθνικών ρυθμίσεων, ανεξαρτήτων εθνικών ρυθμίσεων και θα δημιουργήσει προβλήματα στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Ζητούμε λοιπόν από τον κύριο Μπαρνιέ να θεσπίσει νομοθεσία και έναν κώδικα συμπεριφοράς ε, των χρηστών ούτως ώστε να προστατευθούν οι πολίτες από τον τζόγο στο διαδίκτυο. κύριος Βέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα ότι καλύτερο για την νέα σας θητεία. Τα τυχερά παιχνίδια είναι ένα νέο εθισμό, Ενδεχομένω, μια διαφυγή για τον σύγχρονο άνθρωπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι πλέον γεγονός και επομένω θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο έτσι ώστε να προστατευτούν οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφενό και οι καταναλωτέ αφετέρου. Ποια οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ποια κατεύθυνση. Εάν δώσουμε υπερβολικά μεγάλη αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη, ενδεχομένως θα δημιουργηθούν ε, προβλήματα ε, τα ε, διαδικαστικά και βεβαίως ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κτλ. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να σπάσουν τα μονοπόλια γιατί Ξέρουμε ότι υπάρχουν σε κάποιες χώρες κάποια ε, εθνικά κατά κάποιο τρόπο μονοπόλια, κάποιοι οργανισμοί οποίοι έχουν, στους οποίους έχει δοθεί μονοπωλιακά η δυνατότητα να διαχειρίζονται τα τυχερά παιχνίδια. Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση προς όφελος όλων των πολιτών, των χρηστών ε, ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιγκερέδο για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, εμείς έχουμε ένα θέμα υψίστης της ε, σημασίας για την προστασία των συμφερόντων ε, των λαών και για την καταπολέμηση της απάτης ε, που είναι πολύ συχνές στον, τζόγο, στον τομέα του τζόγου στο διαδίκτυο. Πρέπει τα κράτη να έχουν την αυτονομία τους για να μπορούν να νομοθετούν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ανάλογα με τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε χώρας προστατεύοντας τον καταναλωτή και το λαό τους. Πρόκειται και για επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, όπως γίνεται στην Πορτογαλία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον κανόνα του ελεύθερου ανταγωνισμού και της παροχής υπηρεσιών, διότι δεν πρόκειται για μία παροχή υπηρεσίας. Εδώ πρόκειται για τζόγο που έχει αρνητικά, ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, στους ε, πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί στα κράτη-μέλη όλη η νομιμότητα που έχουν για να νομοθετούν σε αυτόν τον τομέα. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω και να πω δυο λόγια για αυτό το διεθνές πρόβλημα. Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο είναι μεγάλος εθισμός και επομένως Πρόκειται για μια κατάχρηση η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά και άλλα παρελκόμενα προβλήματα στον ε, ε, χρήστη. Ε, ιδιαιτέρως δεν είναι διαδεδομένο αυτό το είδος τυχερού παιχνιδιού ε, στους νέους και επομένως πιστεύω ότι το πρόβλημα θα πρέπει να ξεπεράσει την απλή περιγραφή του και θα πρέπει να περάσουμε στην εξέβρεση λύσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τα γεγονότα, να δούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς συμβαίνει με τα τεχνικά τυχερά παιχνίδια. Ξέρω, ε, ας πούμε, ότι στη δικιά μου μικρή πόλη μέχρι πρώτη υπήρχαν δύο ε, καταστήματα με τέτοια παιχνίδια, τώρα υπάρχουν 18. Θα πρέπει επίσης ε, να καταρτήσουμε τους εκπαιδευτές των παιδιών, τους καθηγητές τους. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος νομίζω, ο κύριος Μόζερ. Σε σχέση με τα online τυχερά παιχνίδια, κατά πόσο πρέπει να διευθύνουν τα μονοπόλια ή θα πρέπει να απαγορευθούν. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε εδώ ότι η αύξηση των εθισμένων στα τυχερά παιχνίδια είναι δραματική. Οι γκρουπιέ στα καζίνο εκπαιδεύονται ε, ούτω ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τους εθισμένους στα τυχερά παιχνίδια και να αποκλείονται από τα καζίνα. Το πρόβλημα του εθισμού βεβαίως τώρα τα καζίνο μετατοπίζεται στο ίντερνετ και με τον τρόπο αυτό διακυβεύεται η υγεία των ε, νέων και συσσωρεύονται χιλιάδες ευρώ σε χρέη. Όσον αφορά την προστασία της νεολαίας, δεν, δεν χρησιμεύει σε τίποτα να απαγορεύσουμε τα τυχερά παιχνίδια. Ένα στους δέκα μαθητές στο Αμβούργο, μεταξύ 15 και 18, παίζει παράνομα με χρήματα, πόκα για παράδειγμα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το κόστος για το, της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και εγώ, γιατί δεν ήμουν παρούσα στην αρχή και επίσης να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για, τις, ε, για τα καλωσορίσματά σας και ευχαριστώ και όλους όσους πήραν το λόγο για την ενθάρρυνση που μου έδωσαν στη νέα θητεία. Όπως γνωρίζετε, το είπα άλλωστε και ενώπιον του Κοινοβουλίου, ότι αυτή η νέα μου θητεία ε, την αναλαμβάνω με μεγάλη αποφασιστικότητα και με λίγη ουτοπία δημιουργική ουτοπία αν θέλετε, ειδικά όταν πρόκειται για τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Όπως είπε και ο, ο πρόεδρος Χάρμπορ ε, πριν από λίγο και όπως είπε και η κυρία Γκέμπχαρτ και ο κύριος Βάρ ε, και ο κύριος Ντεζόγκ ε, με ρώτησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή θα δείξει θέληση, αποφασιστικότητα ε, για να πάρει αποφάσεις και έτσι ώστε να ε, σταματήσουν οποιασδήποτε εσφαλμένες πρακτικές ε, ή οποιοδήποτε παραβιάσει στον τομέα. Αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κατανοήσετε ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να αφήσουμε οτιδήποτε παράνομο να περάσει πολύ μεταξύ μόνο το είπαν και η κυρία Γκέμπχαρτ και ο κύριος Κάρας ε, και πριν από λίγο η κυρία Φιγκερέδο. Δεν πρόκειται για υπηρεσία όπως οι άλλες. Δεν πρόκειται για μια υπηρεσία όπως οι άλλες, το τονίζω και το υπογραμμίζω και έχετε κάθε λόγο να περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα προσέγγιση και μια νέα διαβούλευση την οποία θα σας προτείνω. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ποια θα είναι η προσέγγιση του στο θέμα αυτό αλλά πάντα σε ε, συμφωνία και σε σεβασμό ε, των ε, συνθήκων λαμβάνοντα κυρίω δε υπόψη τον κίνδυνο ε, που ε, επιφέρει για την κοινωνία και για τους νέους ε, ιδιαίτερα ανθρώπους και μάλιστα διάβαζα και την έκθεση της κυρίας Τεμοζέρ και πραγματικά κατανόησα πλήρως το πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές, λέμε, στα κράτη-μέλη. Παρατήρησα ότι από τότε που το 2006 ε, απεφασίστη η απόσυρση του ε, θέματος των χρημάτων από τον κανονισμό για τις υπηρεσίες δεν υπήρξε περαιτέρω διαβούλευση με τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε από πολύ κοντά τις ε, εργασίες της ομάδας του Συμβουλίου που ασχολείται με το θέμα αυτό. Και ξέρω ότι πολλές χώρες μέλη ε, ζητούν ε, τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογή ε, του κανονισμού σχετικά με, τους, με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σας βεβαιώ ότι έχουμε απολύτως, είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία παραβίασης σας βεβαιώ ότι παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά όλο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποβάλλω με προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει διομημένος διάλογος πάνω στο θέμα αυτό. Θέμα το οποίο αφορά έναν νέο ευρωπαϊκού επίπεδου συντονισμό, έναν αποφασιστικό συντονισμό. Και βεβαίω, το θέμα αυτό δεν είναι το μόνο που θα μας απασχολήσει. Υπάρχουν κι άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία αποτελούν πρόκληση γιατί είναι θέματα κοινού ενδιαφέροντος ο κύριος ε, Κυρκόπ ε, και πολλοί άλλοι ε, παρεμβαίνοντες, των οποίων τα ονόματα δεν μπορώ να αναφέρω τώρα, όμως πρέπει να τους πω ότι σημειώνω τα λεγόμενά τους και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι το κύριο διακύβευμα είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Θέλουμε μία ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, που θα αντιμετωπίσει τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ε, δώσουν να έχουμε και κανόνες όσον αφορά ε, το εμπόριο γενικότερα στο διαδίκτυο. Πρόκειται για θέματα τα οποία μελετώνται από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου διότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά και επ' αυτών βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δουλέψει από κοινού με τα κράτη-μέλη. και έστω κι αν κατάλαβα ότι στις διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου μπορεί να εκφράζονται κάποιες διαφορετικές, μερικές φορές και αμφίσιμες ε, απόψεις. Εγώ θα ακούσω όλες τις φωνές του Κοινοβουλίου, όλες τις απόψεις του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης ε, και τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, οργανισμών κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκού επίπεδου διαβούλευση. Αναφέρθηκα σε διακυβεύματα και σε προκλήσεις, κυρία Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω με αυτό. Φυσικά, σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της ε, κοινωνίας ε, το θέμα του εθισμού που αναφέρεται και στην έκθεση ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας ενδιαφέρει και σε σχέση με τους ανήλικες, ανήλικους βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση οι ανήλικοι σε αυτού του είδους τα παιχνίδια και επ' αυτού θα πρέπει να δουλέψουν όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται επομένως ευρωπαϊκό συντονισμός για να ε, δράσουμε σωστά πρέπει να κατανοήσουμε σωστά πρώτα. Και νομίζω ότι το έθιξαν αρκετοί μεταξύ ημών και μάλιστα μερικοί αναφέροντας ε, και ε, αριθμητικά στοιχεία. Και πρέπει να σας πω ότι τα πολιτικά έγγραφα της Επιτροπής περιέχουν και αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία και είναι θέμα το οποίο συζήτησαν και η κυρία Μαγκίνες και άλλοι και πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως το έγγραφο της Επιτροπής ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μονάχα λέξεις, λόγια, ε, αποφάσεις, ε, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μία όσο γίνεται πιο σωστή διάγνωση, έτσι ώστε να βρούμε την όσο γίνεται πιο σωστή λύση. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια είναι το θέμα του αθλητισμού Εγώ ε, ήμουν, είχα την τιμή να είμαι συνδιοργανωτής ε, ε, μεγάλων αγώνων και σε λίγο ξεκινούν και οι Ολυμπιακοί, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί στο Βανκούβερ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία μας και επομένως θα πρέπει να μην αδικήσουμε και αυτές τις διοργανώσεις. Θα ξεκινήσει λοιπόν διαβούλευση και βεβαίως θα γίνει λόγος και για την χρηματοδότηση αθλητικών διοργανώσεων μέσω ε, παιχνιδιών τυχερών ε, ημί. Πρέπει να σας πω ότι πέρα από το Κοινοβούλιο θα έρθω σε επαφή και θα διαβουλευτώ και με άλλους ε, ενδιαφερόμενους και σας ε, ε, βεβαιώ ότι μέχρι το επόμενο φθινόπωρο οπωσδήποτε θα ξαναέρθω μπροστά σας για να σας δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις έχοντας συζητήσει και με τους άλλους επιτρόπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ολοκληρωμένη και ενθαρρυντική απάντηση. Λοιπόν, διακόπτουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπου θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες.